Καλημέρα σε όλους και όλες. Θα μιλήσω στα Σουηδικά. Καλημέρα λοιπόν και στα Σουηδικά. Και καλώς ήρθατε στην σημερινή συνεδρίαση. Μία ανακοίνωση ήθελα να σας κάνω ότι έχουμε αλλάξει την ημερήσια διάταξη λιγάκι. ώστε οι πολιτικές ομάδες να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τον κατάλογο ψηφοφοριών για αύριο. Αύριο έχουμε δύο ώρες ψηφοφοριών. Και έχουμε και την έγκριση της τη διάταξης. Δεν έχω καμία αίτηση για τροποποίηση. Και έχουμε κάποια πράγματα να αλλάξουμε στα πρακτικά. τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων του Δεκεμβρίου, του Νοεμβρίου αλλά και του Οκτωβρίου και έχουμε επίσης έχουμε την, ε, τα πρακτικά των κοινών συνεδριάσεων με άλλες επιτροπές. Εάν δεν έχετε αντίληση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 εξάλληψη της, ε, του γυναικείου ακροτηριασμού των ε, γεννητικών οργάνων. Είναι εμπροετοιμασία το θέμα αυτό και θα έχετε λάβει την ε, τεκμηρίωση και την πρόταση ψηφίσματος. Δεν ήμουν έτοιμος να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι βέβαια σύντομε και συνοπτικέ οι τροπολογίες. Εδώ υπάρχουν τρία θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν ε, αντιμετωπίζουμε την ε, επικείμενη την ε, επικειμένως ανακοινώσιμη πολιτική της Κομισιόν μέσα στο πρόγραμμα της Στοχόλμης που θα έχει και στόχο να αντιμετωπίσει την κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και εδώ θα υπάρχει μια ειδική πρόταση για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, ε, ακροτηριασμών γενικών οργάνων των γυναικών. Η στρατηγική λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς συνδέονται και να λένετε στις διάφορες φορές βίας κατά των γυναικών. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο βασίζεται σε προηγούμενες ε, θέσεις που έχει εκφράσει η Επιτροπή μας. Δεν υπάρχει κάτι το καινοφανές στο κείμενο αυτό και υπάρχει και ένας αριθμός τροπολογιών. Όλα αυτά τα ψηφίσουμε αύριο. Αλλά θα δώσω το λόγο καταρχήν σε όσες και όσους θέλουν. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρούερα. υποστηρίζω αυτό το, αυτή την πρωτοβουλία. Όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά που είπατε και ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό θα γίνει αποδεκτό από αυτούς που πρέπει να το λάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο, <clears throat> σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία είναι αύριο. και εάν όλα πάνε καλά θα πρέπει να έρθει στην πρώτη, στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Προχωρούμε στο σημείο 5. Η απαλλαγή του 2012 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κομισιόν και η κυρία Ματέρα είναι συγγήτρια. Δυστυχώς δεν είναι παρούσα. Αλλά η κυρία Κλάς θα την αντικαταστήσει. Έχετε το λόγο. Καλημέρα. Σας ζητώ να συγχωρήσετε την κυρία Ματέρα, η οποία δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα το πρωί. Μου είπε, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω και να μπορέσω να μεταφέρω τις ε, επιθυμίες της. Πρόκειται για τον, την απαλλαγή για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα των γυναικών. Εδώ πέρα δίνουμε περισσότερη έμφαση στο σημείο 3 και για τα, τις ενέργειες όσοι συγγείται για τα θέματα ενεργειών σε ό,τι αφορά τα θέματα των γυναικών η κυρία Ματέρα εστίασε στο θέμα αυτό της επίτευξης της ισότητας των ε, φύλων. Με αυτήν την ε, γρομοδότηση ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να δώσει έμφαση και να ενσωματώσει το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα θέματα ελέγχου του προϋπολογισμού. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επαναλάβουμε και να γίνει σαφής η θέση μας. Κάνουμε επίσης κάποιες ε, παρατηρήσεις. Λέμε ότι υπήρξε κάποια, υπήρξαν παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου για την αύξηση των σφαλμάτων στην κοινωνική πολιτική και την απασχόληση και φυσικά εκεί πέρα καλύπτονται θέματα ισότητος των φύλων και είναι απαραίτητο να το τονίσουμε αυτό. Θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από, το, από την Κομισιόν στο κατά πόσο αυτές οι, <clears throat> αυτά τα σφάλματα και τα προβλήματα συνδέονται με προγράμματα για την επίτευξη καλύτερης ισότητας των φύλων. Επίσης, προβλέπει αυτή η γνωμοδότηση να υπάρξουν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη περισσότερων στοιχείων και ενδεικτών σε σχέση με την ισότητα των φύλων και να υπάρξει γενική παρακολούθηση και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτής της πολιτικής. Και επίσης η Κομισιόν όταν σχεδιάζει τη χρήση μέσων και κονδυλίων, μέσα λοιπόν στην ε, θέσπιση προτεραιοτήτων και στην απόφαση για τα κονδύλια, ζητείται από την Κομισιόν πάντα να έχει υπόψη της στην οπτική γωνία της ισότητας των φύλων. Και ελπίζω ότι και τα μέλη της Επιτροπής μας θα δεχτούν αυτή τη θέση και αν υπάρχουν περαιτέρω αιτήσει για το θέμα αυτό, είμαι έτοιμη και η κυρία Ματέρα φυσικά να τι αποδεχτεί, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη κυρία Παπαδοπούλου, που δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση για προσωπικού λόγου, θα πω δύο λόγια. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και είμαι σίγουρη ότι θα διαβιβαστεί το μήνυμα. Η κυρία Παπαδοπούλη υποστηρίζει πλήρως τη θέση της εισηγήτριας και επαναλαμβάνει όσοι υπόθηκαν μόλις από τη συνάδελφο ότι είναι κρίμα ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση της εφαρμογής του προπολογισμού της Ένωσης από την σκοπιά της ισότητας των φύλων και δεν γίνεται αναφοράς, ότι αφορά την προώθηση της ισοτροφιλών μέσω των δαπανών και δεν αναφέρονται αυτά στην έκθεση του λεκτικού Συνεδρίου. Πρέπει να ξέρουμε αν ήταν επιτυχή τα προγράμματα και πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα και αν επιτεύθηκαν οι στόχοι και η ανάλυση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της δημοσιονομικής ανάλυσης έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη εξίσου τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών και ότι αξιολογεί το αντίκτυπος των πόρων στους άνδρες και τις γυναίκες και ε, θα πρέπει να βελτιωθούν οι στόχοι των πόρων αν λάβουν υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων ε, και θα βελτιωθεί η συνοχή. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Κομισιόν να ιεραρχήσει με ένα πιο συστηματικό τρόπο θέματα ανισότητα των φύλων στον προγραμματισμό και εφαρμογή όλων των πολιτικών και να διασφαλίσει καλύτερο mainstreaming ε, προκειμένου να πετύχει την πραγματική ισότητα των φύλων. Η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν ε, την υποστήριξη των στόχων ισότητα του φύλου σε ό,τι αφορά ε, τη χρηματοδότηση, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα είναι επίσης ε, κάτι σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι αιτίες, γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζονται για να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες ε, για το θέμα της ισότητας των φύλων και κατάλληλα δεδομένα για να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να προβούμε στην διόρθωση των αρνητικών αποτελεσμάτων και μπορώ να πω ότι για να επιλύσουμε την κρίση χρειαζόμαστε περισσότερη ισότητα και όχι λιγότερη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Μάλιστα. Κανείς δεν το λόγο, οπότε. Μπορούμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών είναι 24 24η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 12 Φεβρουαρίου. Και κατόπιν 17 Μαρτίου και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Και πάλι κυρία Κλάς. Και πάλι θα πρέπει να αντικαταστήσω την κυρία Ματέρα. Ζητείτε εδώ να <clears throat> ζητήσουμε από την Επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού να διερευνήσει τη λειτουργία του mainstream, του gender mainstream, της, ε, προ, της ε, οπτικής γωνίας του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τα θέματα ισότητος των φύλων να εμπλέκεται στο θεσμικό πλαίσιο για τις πολιτικές αυτές. Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει η κυρία Ματέρα ότι οι τρεις λογαριασμοί του Ινστιτούτου που έχουν ένα υπολογισμό 7,7 εκατομμύρια ευρώ απεικονίζουν την δημοσιονομική κατάσταση του Ινστιτούτου και επίσης στη συνέχεια τονίζει ότι το ελεκτικό συνέδριο καταγράφει ότι έχει επιτύχει σημαντικές προόδους το Ίδρυμα αυτό για τις μεταφορές πιστώσεων από το 2012, από το 2011 στο 2012, αλλά παρόλα αυτά για το έτος 2012 έχουν γίνει βελτιώσεις των προσπαθειών για να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση όλων αυτών των ενεργειών. <clears throat> Επίσης, 5η παράγραφο αναφέρεται η παράγραφο αναφέρεται η θέληση του Ινστιτούτου αυτού να εξασφαλίζει τον έλεγχο των πολιτικών και του οργανογράμματος μέσα από ένα πλαίσιο για την εποπτεία του προϋπολογισμού του και στη συνέχεια <clears throat> αναφέρουμε την σημασία της έκθεσης πεπραγμένων του Ινστιτούτου και αναφέρει ότι υπήρξαν δύο εκθέσεις από το Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων και την ε, αλλαγή του κλίματος και έτσι υπήρξε αυτό το έγγραφο το οποίο αποτέλεσε μια σημαντική βάση εργασίας για την για τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η διευθύντρια του Ιδρύματος αυτού ε, έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία και θεωρούμε ότι αυτά μας είναι, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή μας είναι επαρκή για να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να δοθεί η απαλλαγή του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το 2012. Η κυρία Συγγνώμη για την αγνοιά μου, αλλά κάτι δεν πρέπει να κατάλαβα. Δηλαδή θα πάρουν 7,7 ε, εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λαμβάνουν 7,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και τι άλλο κάνουν εκτός από αυτές τις δύο εκθέσεις. Είπατε ότι καταρτίσαν δύο εκθέσεις. Γενικά, θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα όλων αυτών των χρημάτων που δαπανώνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα στη ζωή των γυναικών. Όταν μιλάμε για θύματα, όταν ασκηθεί βία κατά των γυναικών, δεν ε, υπάρχει στην Ουγγαρία, στη χώρα μου, σχεδόν κανένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, πολλά χρήματα δαπανώνται τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γυναίκε δεν βλέπουν τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλω να καταλάβω. Κατάλαβα τα νούμερα, 7,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ότι συντάχθηκαν δύο εκθέσει. Αλλά τι άλλο έχει συμβεί. Σα danke ευχαριστώ και για τις κριτικές παρατηρήσεις σας. Απόλυτα δικαιολογημένα είναι αυτά που λέτε και φυσικά η Επιτροπή μας πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα πάντα να διατυπώσουμε τροπολογίες στις αιτήσεις τους για τα θέματα αυτά. Έχουμε, νομίζω, δεχτεί κατά πλειοψηφία ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας πρέπει να υποστηρίξουν αυτό το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία ελήφθη. Μπορεί να υπάρχουν αιτήσει τροποποίηση σε ορισμένα σημεία και αυτό αφορά και τον προϋπολογισμό και μπορούμε να ζητήσουμε από το Ινστιτούτο αυτό να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο για την πολιτική ισότητα των φύλων. έχει δίκιο η κυρία Μορβάη ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε με κριτικό μάτι την εργασία αυτού του Ινστιτούτου και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την λειτουργία αυτού του Ινστιτούτου. Ίσως θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε την ηγεσία αυτού του Ινστιτούτου για να κάνουμε μια συζήτηση μαζί τους, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο μια συζήτηση για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και αυτό είναι μέσα στα πολιτικά μας καθήκοντα και να τους υποστηρίσουμε αλλά και να ασκούμε πιέσεις προς την κατεύθυνση που μας ενδιαφέρει. Εδώ μας, αναφέρει, μας ενδιαφέρει μονάχα το θέμα της απαλλαγής και τίποτα άλλο. Πριν περάσουμε στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να σας πω ότι στην επόμενη συνεδρίαση Έχουμε προσκαλέσει το Ίδρυμα για την Ισότητα των φίλων ε, για να μας μιλήσει ακριβώς για το έργο του. Θα έχουμε λοιπόν ε, την ευκαιρία, αλλά και στη συνέχεια σήμερα θα έρθει εμπειρογνώμονας από ε, το Ινστιτούτο για την Ισότητα των φίλων και στην επόμενη συνεδρίασή μας θα έρθουν οι διευθυντές του Ινστιτούτου. Και ανά δύο έτη θα έχουμε και μια επίσκεψη προς το Ινστιτούτο αυτό, γιατί βεβαίως και οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Και αυτές οι επισκέψεις είναι ανοιχτές προς όλους. Η ε, κυρία Γκόμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πρέπει και εσείς να το επισκεφτείτε μόνοι σας, γιατί έτσι θα έχετε ε, και μια προσωπική άποψη. Εμεί ε, το επισκεφθήκαμε κατά τη διάρκεια τη Λιθουανική Προεδρία και νομίζω ότι κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύει κανένα εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Δεύτερον, έχουν πολύ μεγάλη βάση δεδομένων ε, για τη διάσταση του φύλου, καλύτερη από την κοινοβουλευτική μελέτη και κάνει πραγματικά πολύ καλό έργο. Αν μελετήσετε προσεκτικά τις εκθέσεις ε, για την ισότητα των φύλων των τελευταίων ετών, θα δείτε την πολυμορφία των προγραμμάτων ε, που έχουν εκπονήσει. βεβαίω το πρόβλημα είναι ότι έχουν ε, πολύ μικρό προσωπικό. Μετά υπήρξαν και οι δημοσιονομικές περικοπές. Τεράστιες περικοπές και στο δικό τους ε, προπολογισμό. Αν πάτε όμως στον ιστότοπο του Ινστιτούτου θα δείτε τι ακριβώς κάνουν, γιατί λειτουργούν με ιδιαίτερα διαφανή τρόπο. Η Διευθύντρια κυρία Λάντπακ πολύ συχνά έρχεται στο Κοινοβούλιο αν υπάρχει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή αν ε, τη χρειάζεται η Επιτροπή μας, πάντα είναι στη διάθεσή μας για να μας βοηθήσει. Όμω και η Νομπορ η Τόμσεν ήταν στην αντιπροσωπεία και βεβαίω ε, και ο πρόεδρο μα ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάτε κι εσεί ε, να δείτε ειδήσει όμω τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι η επίτροπο Ρέντινγκ δεν είχε το χρόνο να πάει κατά τη διάρκεια τη Λιθουανική Προεδρία και αυτό είναι προβληματικό γιατί και εκείνη θα πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει. Καθώ θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει με την ιδιότητά τη γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά. Όμω καλύτερα να πάτε και μόνοι σα για να δείτε τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαβάη. Ευχαριστώ βεβαίως και θα ακούσω με ενδιαφέρον ε, την παρουσίαση αυτών των γυναικών που εκπροσωπούν το Ινστιτούτο σήμερα το απόγευμα, αλλά θα έπρεπε να τονίσω ότι πρόκειται για 7,7 δις ευρώ. Πολύ σημαντικό ποσό εν καιρό κρίσης. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να στηρίξουμε πολλές ε, γυναίκες επιχειρηματίες, να διευκολύνουμε την δραστηριότητά τους, να έχουμε υποδομές για ε, τις γυναίκες που επιβιώνουν από την ε, ενδοκοκοινωνική βία και άλλες μορφές βίας και να καταλάβουμε ότι εμείς που δουλεύουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνηθίσει τέτοια ποσά και δεν μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση τα 7,7 δις. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι Ε, ότι πρέπει να τεκμηρώνονται σωστά αυτές οι επιλογές. Γιατί σε μια διάσταση, αν σκεφτείτε, με το να στηρίξω εγώ αυτή την επιλογή, ε, ουσιαστικά προδίδω την εμπιστοσύνη ε, χιλιάδων γυναικών σε όλη την Ευρώπη που έχουν πολύ που απειλείται η ζωή τους ουσιαστικά. Κύριε ευχαριστώ πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη συζήτηση σύντομα για αυτό το θέμα. Να επενθυμίσω όμω και στη συνάδελφο ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων είναι η έλλειψη δεδομένων. Εναρμονισμένων δεδομένων, μάλιστα. Και ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα από τα κράτη-μέλη για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα πολιτική. Επομένω, πρέπει ακριβώ ε, να παλέψουμε με τα κρατημέλη για να μας δώσουν ε, τα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Αυτό κάνει το Ινστιτούτο και αυτό εμείς στηρίζουμε. Και αν δεν κάνει παραπάνω, είναι επειδή δεν έχει περισσότερες δυνατότητες για να κάνει κάτι παραπάνω. Επομένω, ε, α είμαστε προσεκτικοί πριν τους επικρίνουμε, γιατί ε, παλεύουμε με νύχια και με δόντια να ε, πάρουμε αυτά τα χρήματα και αν δεν τα καταφέρουμε εδώ σε αυτήν την Επιτροπή να πείσουμε τους συναδέλφους, τότε που θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο, και εγώ είχα μπει στο κατάλογο μελητών για αυτό το θέμα. Θα συνεχίσω στο ίδιο μικροσχήματο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ισότητα των φίλων δεν έχουμε αρκετά στατιστικά στοιχεία. για να γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά τα δεδομένα φαίνονται βαρετά ίσως, αλλά αν δεν τα έχουμε στη διάθεσή μας για να εντοπίσουμε τις διαφορές μεταξύ των φύλων, δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από το να καταρτήσουμε, να εκπονήσουμε κάποιες εκθέσεις. Και το Συμβούλιο και η Επιτροπή είχε πολλέ εκθέσει. Έχουν κάνει πολλή δουλειά. Και στο 2013 μάλιστα έθιξαν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τον δίκτυ ισότητας των φύλων. Πρόκειται για ένα δίκτυ που είναι συγκρίσιμος μεταξύ χωρών και μεταξύ διαφορών τομέων. Εστιάζουμε ε, σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας, ε, η επιρροή, η ισχύς και μετά μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων, αν υπάρχει πράγματι ισότητα. Εάν συγκρίνουμε και εξετάσουμε από κοινού όλους, όλα αυτά τα στοιχεία, τότε μπορούμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να συγκρίνω την κατάσταση μεταξύ ε, Σουηδίας ε, και Φιλανδίας. Και γιατί η Δανία, ας πούμε, τα πάει καλύτερα σε έναν τομέα από εμά. Και αυτό αποτελεί τροφή για σκέψη. Ο δείκτης αυτός Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν έχετε 100 σε αυτό το δείκτη, σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη ισότητα. Και μετά μπορείτε να δείτε το μέσο όρο και στα 28 κράτη-μέλη, που είναι 54. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν λοιπόν για να φτάσουμε σε αυτό το 100. Μπορεί βεβαίω να υπάρξει συζήτηση επί του δείκτη, κάποιοι μπορεί να επικρίνουν την ύπαρξη του δείκτη ή τα αποτελέσματα του δείκτη και μετά μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι κρύβεται από πίσω. Ε, με επιστημονικό τρόπο βεβαίω. Το θετικό είναι ότι στην επόμενη συνεδρίαση η Βεγίνα Λάμπακ θα έρθει στην Επιτροπή μας και μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας ε, για να μας πει ακριβώς, ε, να τις πείτε κι εσείς μάλλον, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. Θα είμαστε όλοι εδώ λοιπόν. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Για το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 12 Φεβρουαρίου. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα ψηφίσει στις 18 Μαρτίου και θα περάσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Κλείνουμε αυτό το σημείο. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέρης διάταξης, να σας πω ότι ένα από τα μέλη της Επιτροπής μας απέκτησε παιδί, που είναι κάτι το πάρα πολύ ευχάριστο βεβαίως. Αν κατάλαβα καλά, είχε βάρος 4,3 κιλά το βρέφος, είναι πολύ καλά στην υγεία τους ε, και η μητέρα και το παιδί. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Ξέρουμε αν είναι αγόρι κορίτσι. Όχι. Από βιολογική σκοπιά ήταν κορίτσι πάντως. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2012. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σούμπα, την εισηγητρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα σε σχέση με αυτή την έκθεση να σας πω ότι πιστεύω ότι η συνεργασία η οποία έχει γίνει μεταξύ των σκυριωδών συγητών, έχει καταλήξει σε συμβαστικέ λύσει, οι οποίε μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ικανοποιητικέ για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση. Ήταν αρκετά ε, πλούσια η εργασία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτό. Έχουμε πάνω από 20 συμβιβαστικές τροπολογίες που έτυχαν συμφωνίας. Ήταν όλα αυτά λοιπόν ιδιαίτερα θετικά Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες θα μπορέσουν να υποστηριχθούν από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες εστιάζουν σε δύο ή τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο από αυτά τα ερωτήματα έχει να κάνει φυσικά με την ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας και πολιτικής που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τον τρόπο αυτή η κατάσταση έχει άμεσες επιπτώσεις, ειδικά στις γυναίκες, επειδή βλέπουμε να μειώνεται η ισότητα, να μην επιτυγχάνεται η ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών λόγω και της κρίσης. Επίσης, βλέπουμε να συνεχίζεται με την οικονομική κρίση η διαιώνιση της ανισότητας ανδρών και γυναικών και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία έχουν αναλυφθεί για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και Προφανώς αυτά τα μέτρα δεν είναι σαφές ότι είχαν πάντα τις απαραίτητες πρόνοιες για να αντιμετωπιστεί η επίτευξη της ισότητας ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε ορισμένε κοινέ θέσεις που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά θέματα, με τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας, με την διαφορά των εργασιακών συνθηκών μεταξύ ανδρών και γυναικών, με την διαφορά απολαβών οικονομικών και αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τις διαφορές σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές και τα λοιπά. Άλλες συμβαστικές τροπολογίες έχουν να κάνουν με τις ανησυχίες για τα θέματα βίας κατά των γυναικών, για την ε, εμπορία γυναικών και επίσης αναφερόμαστε στις, στις ποσοστώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της επισφαλούς εργασίας για τις νέες γυναίκες. Καταφέραμε λοιπόν για να, να καλύψουμε τις πάνω από 300 τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβασικές τροπολογίες. Πρέπει επίσης να πω ότι στις ε, εκτιμήσεις μου που απεικονίζονται στην ε, λίστα ψηφοφοριών για τις περισσότερες τροπολογίες εγώ υποστηρίζω την ψήφισή τους. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα για τα οποία έχω ακόμα κάποιες αμφιβολίες και αυτό φαίνεται και στην αξιολόγησή μου. Για την τροπολογία τώρα 170 που έχει κατατεθεί από την κυρία Μπέρες έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το περιεχόμενο και το νόημα αυτής της τροπολογίας. Το θέμα εκεί ήταν τα θέματα των συμβάσεων εργασίας και η δική μου πρόταση ήταν η κάθε μόνιμη θέση εργασίας θα πρέπει να καλύπτεται από, ένα, από μια ουσιαστική σύμβαση εργασίας Και η τροπολογία εδώ λέει ότι όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να καλύπτονται από μια αποτελεσματικού χαρακτήρα σύμβαση. Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι μια καλή και θετική πρόθεση, πιστεύουμε ότι σε επίπεδο ρεαλιστικό δεν μπορούν όλες οι θέσεις εργασίας να είναι θέσεις εργασίας που έχουν μόνιμο και ε, πραγματικό χαρακτήρα, γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις εργασιακές συνθήκες, είναι απαραίτητο πολλές φορές να καλύπτονται ανάγκες σε προσωρινό επίπεδο και όχι με μόνιμα συμβόλαια. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε περισσότερο μαζί με τους σοσιαλιστές ή με την ίδια την κυρία Μπερές, η οποία πρότεινε αυτή την τροπολογία. Και επίσης για τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν να κάνουν τις ποσοστώσεις και για την είσοδο των γυναικών βάσει ποσοστώσεων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η δική μου θέση για το θέμα αυτό δεν είναι ευνοϊκή. Γιατί και εγώ προσωπικά και το κόμμα μου έχουμε μια πολιτική θέση σε σχέση με τις ποσοστώσεις. Θεωρούμε ότι οι ποσοστώσεις αυτές δεν επιλύουν το ουσιαστικό πρόβλημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά, και αυτό είναι δική μου θέση, με την οποία δεν θα συμφωνήσουν ίσως πολλοί βουλευτές από τη δική μου πολιτική ομάδα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στη ψηφοφορία Ε, η πολιτική μου ομάδα φυσικά έχει πολυπίκυλες απόψεις για το θέμα αυτό. Αυτά τα οποία εγώ λέω λοιπόν είναι η θέση του δικού μου κόμματος και η δική μου. και πιστεύω ότι το θέμα των ποσοστώσεων δεν είναι ένα θεμελιώδης θέμα για το οποίο εμείς θα πρέπει να εκφέρουμε γνώμη Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να εστιάσουμε υπερβολικά σε αυτό το θέμα, στη συγκεκριμένη αυτή την έκθεση και δεδομένου ότι δεν έχουμε κοινέ απόψεις σε όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ότι ε, υπάρχει γενικά για τα υπόλοιπα θέματα μία συγκλίνουσα άποψη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς και όλες αυτές οι οποίες συνεργάστηκαν μαζί μου για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτές τις ε, συμβιβαστικέ προτάσεις τροπολογιών που είναι πια σε τελειωτική σχεδόν μορφή. Θέλω να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες, τις σκιώδεις εισηγήτριες και τη γραμματεία, ιδιω την Άντζελα, η οποία κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να περατωθούν αυτές τις εργασίες. Ευχαριστούμε. Eh, Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε ποιον τον επιθυμεί. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Χάνιμπολ. Ναι, ευχαριστώ. Έχω μια δήλωση από την κυρία ε, και θέλω ε, και εγώ ε, να αναφερθώ στη γέννηση του μωρού και όλοι στέλνουμε τα συγχαρητηριά μας, ε, Άννα νομίζω λέγεται το μωρό. Η κυρία Κλαβακέκους θα ήθελε καταρχήν να συγχαρεί την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της πιστεύει ότι όλα τα κυρία σημεία έχουν συμπεριληφθεί στις τροπολογίες και στις συμβαστικές τροπολογίες ε, και η κυρία Χρυβακάκους ε, υποστηρίζει πλήρως ε, τις τροπολογίες που αναφέρονται στα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας στις γυναίκες. Εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα και αυτό επηρεάζει τις γυναίκες και υπάρχει και χάσμα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Επίσης αναφέρεται και στο πρόβλημα της Φιλίωσης της ε, οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Χρειαζόμαστε ε, καλύτερες ε, υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών ε, και πρέπει να υπάρξει υποστήριξη των γυναικών για να μπορούν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να μπορούν να βρουν μόνιμες δουλειές με πλήρη επιδόματα. Επίσης αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών που αυξήθηκε με την κρίση. Χρειαζόμαστε καλύτερη παροχή συμβουλή και πιο φθηνή για τα θύματα. Και θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα ε, της ε, ασφάλειας ε, των θέσεων εργασίας και των συμβάσεων και στις απόψεις της κυρίας Μπερές. Η δική μου ομάδα και εγώ θα υπερασπίζαμε να έχουν όλοι μια κανονική σύμβαση εργασία, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε είμαστε ευάλωτοι σε πολλά. Το υποστηρίζω λοιπόν αυτό και το άλλο θέμα για τι ποσοστώσει ε, για τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Έχει περάσει η πρόταση αυτή και η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υποστήριξε το θέμα αυτό πάρα πολύ και εγώ έχω έντονες απόψεις γι' αυτό, αν και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ίσως μπορεί να μην επιληθούν κάποια από τα κύρια προβλήματα της ενισότητας, είναι ένας ε, τρόπος ε, και αυτός και όταν ε, κάποιες γυναίκες, όταν οι γυναίκες καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις διευθύνουσες, τότε αυτό γίνεται πιο αποδεκτό και στη δική σας ε, χώρα, Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει, πάει πολύ καλά η χώρα σας αυτό και έχει περισσότερες γυναίκες τώρα στο Κοινοβουλίο, νομίζω, από ότι άντρε. Επομένως, είδαμε αποτελέσματα και νομίζω ότι αν το υθετήσουμε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δούμε τα ίδια αποτελέσματα και το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλβάου Μπαραντίκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έκανε για να προετοιμάσει τις συμβαστικές τροπολογίες που μας παρουσίασε η δική μας ομάδα συμφωνεί με τις συμβαστικές τροπολογίες που συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και όπως είπαμε και στην πρώτη συζήτηση, η ε, το σχέδιο βασιζόταν σε οικονομικές πτυχές για το θέμα της προσέγγισης της ισότητας και εμείς ε, θεωρήσαμε ότι ε, πρέπει και οι δημόσιες πολιτικές ε, να προσμετρήσουν τη συνεισφορά των γυναικών στην ευημερία και στην οικονομική ανάπτυξη και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μέσω της δουλειάς τους που ε, δεν πληρώνεται δεν αποζημιώνεται. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η προσπάθεια ε, για να αξιολογηθεί αυτή η συνεισφορά για να δοθεί και μια διαφορετική προοπτική. Επίσης δεν θα πετύχουμε την ισότητα αν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική ευέλικτων ωραρίων έτσι ώστε να μπορεί να ε, προσαρμόζεται η κάθε οικογένεια ανάλογα με τις ανάγκες της. Ήταν επίσης απαραίτητο να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα δεδομένη τη οικονομική κατάσταση και δεδομένη τη πραγματικότητα των συμβάσεων, ήταν απαραίτητο να ενσωματώσουμε με δημόσιε πολιτικέ τι γυναίκε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, όχι μόνο λόγω. Ε, εξαιτία του ότι είναι αυτοδίκαιο, αλλά και λόγω ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα που μα δείχνουν ότι αν οι γυναίκε ε, συμμετέχουν ε, σε περιβάλλοντα ε, εργασίας, τότε επιφέρουν περισσότερη ανταγωνιστικότητα, περισσότερη δημιουργικότητα και βελτιώνουν και τα οικονομικά των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις στιγμές κρίσης δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για αρνητικά πράγματα και για επισφάλεια, αλλά και για προτάσεις που θα μας πάνε μπροστά. Επίσης, δεν θα προχωρήσουμε στο θέμα της ισότητας αν δεν εργαστούμε για την εξάλληψη των στερεοτύπων που τα βλέπουμε συνεχώς, αλλά και εδώ, καθημερινά και σε αυτό το κοινοβούλιο, δηλαδή και στη γλώσσα ε, και στις εικόνες και στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν εγκάρσιο χαρακτήρα και θα πρέπει να επιμένουμε σε αυτά τα θέματα σε όλες τις εκθέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν οι διαπραγματοί τροπολογίες μας και να σας πω ότι ναι, αποφασιστικά πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ πρέπει να πω ότι πριν 20 ε, χρόνια εγώ δεν ήμουν και τόσο υπέρ των γιατί έλεγα ότι ε, θα ενταχθούμε για οι γυναίκες ε, αφού σπουδάζουμε, όμως είδα ότι τελικά δεν υλοποιείται κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν θα πω ναι και θυμάμαι τι μου είπε μια φίλη μου στη συζήτηση αυτή και μου είπε και εσύ γιατί θέλεις ε, να έχουμε αυτές τις ποσοστώσεις. Εγώ ε, είπα ότι θέλω κάτι τέτοιο για να μπορούμε και εμείς ε, να κάνουμε τόσα λάθη όσο και οι άντρες. Και εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της, για την εξέβρεση συμβασμών. Το ΕΛΚ βεβαίω θα τι υποστηρίξει όλε, όμω θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήταν επικοδομητική συνεργασία μα και το έργο τη ηγήτρια και βεβαίω θα υπάρξουν και free votes ε, για τι ε, ποσοστώσει και άλλα θέματα. Τώρα, για το ίδιο το προσχέδιο, το ΕΛΚ και εγώ η ίδια έχουμε καταθέσει πάνω από το 1 τρίτο των ε, τροπολογιών. Να θυμίσω ότι δεν ήταν εύκολο το έργο τη εισηγήτριας. Όμως, θεωρούμε ότι το προσχέδιο ήταν, ε, εστίαζε ιδιαίτερα ε, στην οικονομία, αλλά ήταν και αρκετά απεσιόδοξο και γενικευμένο. Για παράδειγμα, τα μέτρα λιτότητα, με ιδιαίτερα γενικευμένο τρόπο και δυσανάλογο κάποιες φορές, ε, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα σύνδεση με τις ανισότητες, δεν αντικατόπτριζε την πραγματικότητα και στα 28 κράτη-μέλη, εφόσον θεωρείται ότι θα υπάρχουν και ανισότητε και κάποιε διαφορέ ήταν εξαιρετικά σημαντικό να, να επενθυμίσουμε ότι μπορεί και εθελοντικά γυναίκες να θέλουν να δουλέψουν ε, ε, με ευέλικτους όρους εργασίας, ε, με μερική απασχόληση. Και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα κακό, όπως επίσης θα πρέπει να μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο τομέα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ε, δηλώσεις που μας ε, φαίνονται ιδιαίτερα ιδεολογικές. Πέραν της ε, μισθολογικής ισότητας και της απασχόλησης, εδώ θέλουμε να εξετάσουμε με σφαιρικό τρόπο την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων για το 2012. Έχουμε καταθέσει λοιπόν 124 τροπολογίες. Ε, πρώτον υπενθυμίζουμε και πάλι στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαϊκέ οδηγίε για την ε, ίση μεταχείριση ανθρώπων και γυναικών θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει και είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο επίση είναι να συνεχίζουμε ε, το χάσμα το μισθολογικό, αλλά για το 2012, παρά την κρίση και στην απασχόληση, θα πρέπει να ε, δούμε ακριβώς τι είδαμε, τι παρατηρήσαμε, ότι το χάσμα μειώθηκε ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών από την κρίση, γιατί ε, κυρίως επλήγησαν οι τομείς απασχόλησης των ανδρών. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ότι δεν... οι γυναίκες δεν είναι θύματα και διαρθρωτικών ανισοτήτων. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Εκεί βεβαίως δεν υπάρχει πρόοδος. Επιμένουμε στη σημασία της προώθησης κάποιων επαγγελμάτων στις γυναίκες, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των ε, κοριτσιών, των γυναικών, στους ε, τομείς που αναπτύσσονται και εκεί όπου υπάρχουν κάποια εχέγγυα ίσων απολαβών. Να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη που θα διασφαλίζουν κατά τη διάρκεια των ε, σπουδών οι νέοι άντρε και οι νέε γυναίκε, θα έχουν τις ίδιες ε, ευκαιρίες και προοπτικές που δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται τώρα. Πρέπει να θεωρήνουμε και τους ε, εργοδότες αυτών των τομέων να επιλέγουν περισσότερο τις γυναίκες, για παράδειγμα στον εμπορικό κόσμο. Υπήρξαν και αντίστοιχε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που μας ε, βοήθησαν. Τώρα, υπογραμμίζουμε τη σημασία λήψης συγκεκριμένων μέτρων για να υπάρξει καλύτερος καταμορισμός των ε, καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την οικογένεια, για την απασχόληση και το καθεξής. Βεβαίω αυτό δεν είναι μόνο θέμα δημόσιας πολιτικής, κάτι το οποίο υπονοείται στο προσχέδιο, αλλά και στην δέσμευση και συμβολή των εργοδοτών και των επιχειρήσεων. Μια τροπολογία που θεωρώ σημαντική, και εδώ βεβαίω υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, είναι το λεγόμενο family caregiver status, που αναγνωρίζει ε, τις γυναίκες ε, που ε, στηρίζουν τους συγγενείς τους, για παράδειγμα, αλλά και νομιμοποιεί και αναγνωρίζει το ρόλο και το, τη σημαντική του συμβολή στην κοινωνία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης και την, το ιδιαίτερο ευάλωτο της κατάστασης κάποιων γυναικών που αντιμετωπίζουν αναπηρίαση ή έχουν παιδί με αναπηρία. Για τα στερεότυπα Καλούμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν περισσότερα προγράμματα ευαισθητοποίηση ε, για ε, τους εφήβους, να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα σε ό,τι αφορά την ε, εικόνα της γυναίκας στον τύπο. Μετά τέλος για την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό και στις επερχόμενε εκλογές, αλλά και για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Επιμένουμε στο γεγονό ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η ισότητα των ε, φύλων στη νέα επιτροπή που θα διαμορφωθεί. Ελπίζουμε αυτό να συμβεί και έχουμε καταθέσει και τροπολογίε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση ε, τη βία κατά των γυναικών. Στηρίζουμε και την ιδέα τη Παρβένοβα και άλλων το 2016 να αφιερωθεί στην καταπολέμηση τη ε, βία κατά των γυναικών. Και ξέρω ότι η κυρία Ζουμπέρ, εντάξει, δεν ε, θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχουν ποσοστώσει. Σα προσκαλώ να έρθετε στο Βέλιο και να δείτε πραγματικά πόσο καλά λειτουργεί αυτό το σύστημα. Θα δείτε τα στοιχεία και θα δείτε ότι αυτό λειτουργεί σε εμά. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, είχαμε πολλέ τροπολογίε. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος. Θέλει να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ξαναδίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ. Στην ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, εγώ ήδη ανέφερα το γεγονός ότι η έμφαση επί των οικονομικών θεμάτων κατά την άποψή μου, αιτιολογείται αν λάβουμε υπόψη τη συγκυρία στην οποία ζούμε, αλλά ανεξάρτητα από τη δική μου προσωπική άποψη. Είναι σημαντικό να ξαναθυμίσουμε ότι αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί βάσει της αξιολόγησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων το 2012 και αυτή η αξιολόγηση της Κομισιόν εστιάζεται ουσιαστικά, εστιάζει ουσιαστικά σε οικονομικά ζητήματα και αυτή η ολόγηση δεν είναι δική μου αλλά της Κομισιόν ότι αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά ως προς τον αντίκτυπο που έχουν σε θέματα ισότητας. Ε, έτσι λοιπόν, αυτά παρουσιάστηκαν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πρέπει να πω ότι το βάρος που δίνεται στην έκθεση στα θέματα αυτά αντικατοπτρίζει <laughs> απλώς την προτεραιότητα που έδωσε η ίδια η Κομισιόν στα στοιχεία και στην αξιολόγηση που παρουσίασε για το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων το 2012. Ένα από τα θέματα που επίσης θεωρώ σημαντικά να διευκρινίσω και είναι αρκετά επίμαχο είναι το θέμα της ε, εργασίας, της μερικής απασχόλησης και του χαρακτήρα αυτού του είδους της εργασίας, ε, δηλαδή αν μιλάμε για εθελοντικό ή μη εθελοντικό χαρακτήρα. Κατά τη δική μας άποψη και έχοντας κατά νου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, οι εργοδότες είναι αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούν στις αναγκαιότητες των γυναικών. Εμείς λοιπόν θέλουμε να θέσουμε αυτό τον εθελοντικό χαρακτήρα αυτού του είδους εργασίας, γιατί αν δεν το κάναμε, Ομόμαστε ότι θα υπήρχε χειραγώγηση αυτής της αναγκαιότητας των γυναικών ενίοτε να έχουν μερική απασχόληση. Είναι προφανές ότι Έχουμε διαφορετικές πραγματικότητες ε, στο διάφορα κράτη-μέλη και εγώ βασικά γνωρίζω περισσότερο την πραγματικότητα της Πορτογαλίας όμως. Στις ε, χώρες αυτές ε, ξέρω ότι οι σύμβασεις μερικής απασχόλησης, κυρίως απευθύνουν στις γυναίκες και και πολλές φορές αμείβονται με 250-300 ευρώ. Και δεν θέλουν φυσικά κάτι τέτοιο οι γυναίκε, αλλά πρέπει να το δεκτούν γιατί δεν έχουν εναλλακτική. Και προφανώ. κάτι τέτοιο δεν ε, εγγυάται την οικονομική ανεξαρτησία κανενός ε, και πόσο μάλλον των γυναικών. Επομένως, η ανησυχία μας εδώ είναι να εγγυθούμε ότι τέτοιου είδους εργασία, ναι πρέπει να υπάρχει, πρέπει να μπορεί να υπάρχει, αλλά θέλουμε να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες των γυναικών, στις ανάγκες των γυναικών. Δεν θέλω τώρα να προκαλέσω εδώ πολεμική. Όμως θέλω να πω ότι θεωρώ σημαντικό οι γυναίκες που ποινικοποιούνται επειδή έχουν άτομα να αυτές, να ε, αναγνωρίζετε η αξία τους, να μην ζημιώνονται από τους άλλους, αλλά επίσης δεν θα ήθελα να εδρεωθεί εδώ η ιδέα ότι το ρόλο αυτό τον έχουν γυναίκες και είναι ένας ρόλος φυσικός οι τροπολογίες, κάποιες τροπολογίες ε, που συντάχθηκαν δεν πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση να εγγυηθούν οι γυναίκες που ασκούν αυτού του είδους την εργασία να μην ζημιώνονται επειδή δίνουν αυτή τη βοήθεια που είναι τόσο απαραίτητη. Και ξέρουμε ότι σήμερα στις κοινωνίες μας ε, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια που να υποστηρίζει τις οικογένειες στα ζητήματα αυτά. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία όπως ξέρετε για το ζήτημα αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει στην Ολομέλεια το Μάρτιο, εάν θέλει και ο Θεός. Θα είναι μακρά η ψηφοφορία, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για αυτή την έκθεση. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο ε, σημείο 8, που είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση της πορνείας και η επίπτωσή της στην ε, ισότητα των φύλων θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάνιμπαλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένιωσα μεγάλη χαρά και τιμή που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την έκθεση για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και γίνεται όλο και πιο σημαντικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ένα θέμα που σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά τις γυναίκες, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην πορνεία είναι γυναίκες, 99% συγκεκριμένα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν θέμα για την Επιτροπή μας και ένα θέμα που έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα. Χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Η ελπίδα μου είναι ότι θα γίνει δεκτή αυτή η έκθεση και θα μπορέσει να φτάσει στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τις πολιτικές τους και την νομοθεσία που ισχύει σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η, προ... η πορνεία στρέφεται από τη βάση της κατά της ισότητας των φύλων. Είναι μια άνηση συμφωνία που επιτρέπει στους άνδρες να αγοράζουν τα κορμιά των γυναικών. Μπορεί να είναι το παλιότερο επάγγελμα και να υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτός δεν είναι κανένας λόγος για να συνεχίσει να ισχύει για χιλιάδες χρόνια. Είναι κάτι που στρέφεται εναντίον των γυναικών και, αυτή είναι, και αυτός είναι ο κύριος άξονας της έκθεσής μου. Δεν είμαι τόσο ιδεαλιστική <clears throat> ώστε να πιστεύω ότι αύριο μπορεί να εξαλειφθεί η πορνεία ή σε λίγα χρόνια. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να εισαγάγουμε μέτρα τα οποία θα μειώσουν την πορνεία και τις εγκληματικές δραστηριότητες που την περιστοιχίζουν. Αυτή είναι η ελπίδα μου με την έκθεση αυτή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει και το αναφέρω στην έκθεση ότι οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό ακριβώ κάνει η πορνεία. Η πορνεία με ευρύτερη έννοια είναι κάτι το οποίο στρέφεται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά στην Επιτροπή μας, υπήρξαν πολλές προσεγγίσεις στα θέματα της πορνείας. Και όλα αυτά καλύπτουν διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Υπάρχει η άποψη που έχω αναφέρει εγώ προηγουμένως και που πιστεύω πρέπει να είναι η βάση της δικής μας ανάλυσης ότι η πορνεία ε, την ισότητα των φίλων και στρέφεται κατά των γυναικών. Υπάρχει όμως και μία άποψη η οποία είναι έγκυρη από εσμένε ε, πλευρές αλλά δεν εφαρμόζεται επιτυχώς στην πράξη είναι ότι οι γυναίκε θα πρέπει να είναι ελεύθερε να διαθέσουν όπω θέλουν το σώμα του. Κάτι το οποίο είναι έγκυρο μέχρι ένα σημείο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι οι γυναίκε γίνονται πόρνε επειδή θέλουν να διαθέτουν ελεύθερα το σώμα του. Είχα πολλέ συζητήσει με εργαζόμενου του τομέα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ υψηλό βαθμό λαθρεμπορία γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κομισιόν έχει στοιχεία τα οποία και ξέρω ότι είναι δύσκολη συλλογή στοιχείων, αλλά τα στοιχεία των, ε, που έχει συλλέξει η Κομισιόν λένε ότι 80% των γυναικών που είναι στην πορνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τύχη λαθρεμπορίας γυναικών και επίσης υπάρχει και η εγκληματική οργάνωση που έχει να κάνει με την πορνεία που φέρνει σημαντικά ε, κέρδη στον υπόκοσμο και βρίσκονται στη δεύτερη θέση μόνο μετά από το εμπόριο ναρκωτικών. Ακόμα και στις χώρες που όπου είναι νόμιμη η πορνεία. Η νομοποίηση της πορνείας δεν εμποδίζει τις εγκληματικές ενέργειες που κρύβονται πίσω από την πορνεία. Ακριβώς επειδή είναι ε, νομιμοποιημένη η πορνεία σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία είναι περισσότερος ο όγκος των δραστηριοτήτων και αυτό γεννά περισσότερες εγκληματικές ε, ε δραστηριότητες. Στην ε, Ολλανδία, στη Γερμανία και την Ελλάδα είναι νόμιμη η πορνεία, σε άλλες χώρες δεν είναι νόμιμη, αλλά ποινικοποιούνται οι ίδιες οι πόρνες. Αυτό συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η... δεν είναι παράνομη η πορνεία, αλλά η προσέλκυση πελατών ή η λειτουργία ενός ε, Πορνίου είναι κάτι το οποίο είναι μια παράνομη διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και στην Ιρλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου ισχύει ένας αντίστοιχος νόμος και όπου ποινικοποιούνται όχι ε, μονάχα οι πελάτες αλλά και οι πόρνες. Το άλλο μοντέλο το οποίο κερδίζει όλο περισσότερη υποστήριξη είναι το σουηδικό μοντέλο το οποίο ισχύει και στην Νορβηγία και την Ισλανδία. Η Σουηδία φυσικά είναι η μόνη χώρα η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι ο αγοραστής σεξουαλικών υπηρεσιών ο οποίος θα πρέπει να κολλάζεται. Έχει ποινική ευθύνη. Είναι οι άνδρες λοιπόν οι οποίοι αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες που είναι ένοχοι ποινικών ε, αδικημάτων. Υπάρχουν πολύ έντονα στοιχεία από τη Σουηδία που καταδεικνύουν ότι αυτό έχει μειώσει την πορνεία και έχει αλλάξει την αντιμετώπιση προς τις ε, πόρνες και τα νέα κορίτσια βλέπουν ότι η πορνεία είναι μια δραστηριότητα στην οποία δεν θέλουν να εμπλακούν και είναι εναντίον αυτής. Είναι πολλά τα θετικά λοιπόν αυτού του μοντέλου και στη Γαλλία όπου η κατάσταση ήταν παρόμοια με αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου και ακολουθεί να είναι, τώρα περνάει από το Γαλλικό ε, Κοινοβούλιο, από τη Γερουσία συγκεκριμένα έχει περάσει από την ε, Βουλή των Αντιπροσώπων που εφαρμοζεί το σουηδικό μοντέλο και ποινικοποιεί τον αγοραστή σεξουαλικών υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι λοιπόν, ένα μοντέλο το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξιοπιστία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου μοντέλου θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο γιατί οι γυναίκες μπαίνουν στον χώρο της πορνείας. Δεν νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ελεύθερη επιλογή. Πολύ λίγες γυναίκες είναι, αυ... αυτές οι οποίες το κάνουν εθελοντικά, παρά το γεγονός ότι τα λόμπι των ε, των εργαζομένων σε αυτό το τομέα θέλουν να δώσουν αυτή την εντύπωση. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως σας είπα προηγουμένως, δείχνουν ότι πάνω από 80% των εργαζομένων στην πορνεία είναι θύματα βίας, ε, ε, βιασμού, αιμομιξίας, παιδοφιλίας και αυτό τις έχει οθήσει στην ε, πορνεία. Κάποιες μπορεί να το κάνουν για οικονομικούς λόγους, αλλά σχεδόν ποτέ δεν είναι αυτό μια ελεύθερη επιλογή. Αν μια γυναίκα πηγαίνει στον χώρο της πορνείας επειδή είναι θύμα σεξουαλικής βίας ή επειδή δεν έχει καμία άλλη διέξοδο για να υποστηρίξει την οικογένειά της, δεν μιλάμε για μια ελεύθερη επιλογή, δεν είναι αποφάσεις που πηγάζουν από τη θέληση να ακολουθήσει κανεί ένα επαγγελματικό τομέα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια απασχόληση όπω οποιαδήποτε άλλη η πορνεία. Και εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν καταλαβαίνω αυτούς που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι καμία γυναίκα, κανένα μέλος αυτής της Επιτροπής που θα έλεγε εθελοντικά εντάξει από αύριο θα αρχίσω να εκπορνεύομαι. Αν υπάρχει κάποια η οποία έχει διαφορετική άποψη να μας το πείτε και αν δεν θέλετε να το πείτε δημόσια πείτε το ιδιωτικά σε μένα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τις γυναίκες και για την ισότητα των φίλων και η έκθεσή μου τονίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το σουηδικό μοντέλο και ίσως αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός. Η ελπίδα μου λοιπόν είναι ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε την έκθεσή μου. Έκανα πολλές συζητήσεις με τις σκιώδεις εισηγήτριες που με υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν την κατεύθυνση αυτή. Υπήρξε μια επικοδομητική συζήτηση για τα θέματα αυτά και όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια έκθεση που ελπίζω ότι όλοι και όλες μας μπορούμε να υποστηρίξουμε γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις γυναίκες και είναι κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο. Κυρία Δουβή. My micro. Oh, Εντάξει, λειτουργεί το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που υπάρχει διερμηνία προς τα εστονικά. Μπορώ να μιλήσω έτσι τη μητρική μου. Ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Χάνιμπολ για το έργο της και να ευχαριστήσω όλους όσοι κατέθεσαν τροπολογίες. Το 85% ημών έχει την ίδια στάση απέναντι στην πορνεία. Είμαστε κατά της πώληση του ίδιου μας του κορμιού οι τροπολογίες μας παρουσιάζουν δύο προσεγγίσεις προς την πορνεία. Τις ανέφερε και η κυρία Χόνιμπολ. Η μία προσέγγιση υποστηρίζει την ποινικοποίηση της πορνείας. Είναι η κυρίαρχη επιλογή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην οικονομία της αγοράς, αν δεν υπάρχει ζήτηση δεν μπορεί να υπάρξει προσφορά, ενώ από την άλλη το σοηδικό μοντέλο είναι πολύ καλό, όλοι θα έπρεπε να το ακολουθήσουμε. Και υπάρχει και άλλη μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το σώμα τους. Δεν θέλω να αναφερθώ στους λόγους ε, για τους οποίους το 98% των ε, γυναικών που εργάζονται ως πόρνες ε, έχουν επιλέξει αυτό το δρόμο. Αλλά μελέτες και αναλύσεις δείχνουν ότι αυτοί οι λόγοι δεν έχουν καμία σχέση με τη λεγόμενη ελεύθερη επιλογή. Προ εκείνου τους πολιτικούς ε, που υποστηρίζουν την εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος, θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση δεν απαγορεύει το ελεύθερο συνενετικό σεξ. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί να επιτρέψουμε την πορνεία και όλες τις, τις επιπτώσεις, το οργανωμένο έγκλημα και το καθεξής. Είμαι πεπισμένη ότι η ποινικοποίηση των σεξουαλικών υπηρεσιών, της πορνείας, θα ωφελούσε την κοινωνία. Γιατί έτσι θα μειώνονταν τα τραβάσανα χιλιάδων ανθρώπων, αν δεν υπήρχε πορνεία. Έχω μία ακόμα παρατήρηση πέραν της ε, ποινικοποίησης της πορνείας. Στην έκθεση αυτή και στις τροπολογίες ε, έχουμε μπερδέψει τον όρο κορίτσι και ανήλικο άτομο. Τι εννοούμε κορίτσι εδώ. Μάλλον εδώ εννοούμε ανήλικη και δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε να πούμε ξεκάθαρα ότι η πορνεία ανηλίκων είναι κάτι το εντελώ απαράδεκτο. Το κορίτσι δεν είναι νομικός όρος. Μιλάμε για μια κοπέλα που είναι 19 με 21. Τι ακριβώς εννοούμε εδώ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τους ε, όρους ε, που χρησιμοποιούμε και να υπάρξει και εναρμόνιση από πλευρά τη εισηγήτρια. Στην σύμβαση ε, για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ αναφέρεται ότι το παιδί είναι οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Το ανήλικο άτομο είναι ο μόνος νομικός όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω μόνο στο εξή. Πρόσφατα άκουσα ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί των παιδιών ή των κοριτσιών. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, το κορίτσι, ως κορίτσι ορίζεται οποιοδήποτε κορίτσι κάτω των 18. Βεβαίω μπορεί να υπάρχουν διαφορές, αλλά για μένα το κορίτσι είναι παιδί, είναι ανήλικο. Παρακαλώ. Αν και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορέ. Ναι. Μια σύντομη παρατηρήση. Αν εξετάσετε το διεθνέ δίκαιο, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, που είναι από τα πολύ βασικά κείμενα όταν εξετάζουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Εκεί ω παιδί ορίζουμε ένα ανήλικο άτομο κάτω των 18 ετών. Όταν μιλάμε για κορίτσια, Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι εννοούμε και τις νέες γυναίκες ε, ηλικίας 19 έως 21 ετών, για παράδειγμα. Αλλά το παιδί, όρος παιδί, είναι περισσότερο συναισθηματικός παρά νομικός όρος. Εντάξει, ωραία, σε συνεχίσουμε. Η κυρία Μόρβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μ' ακούτε τώρα, ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερως που έχουμε αυτή την έκθεση και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση, αλλά και όλους ε, όσοι εργάστηκαν από αυτής. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά αυτή την ε, αλλαγή που γίνεται ε, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που ακολουθούμε μετά από αυτή την έκθεση. Πρώτον, από ιστορική σκοπιά η κοινωνία πάντα θεωρούσε τη γυναίκα ως ε, τον μοναδικό φορέα σφαλμάτων Πάντα έτσι βλέπαμε τις γυναίκες ως τις μόνες που σφάλουν. Ε, αυτό το είδαμε και πιο πρόσφατα με, την, ε, με τις εκτρώσεις. Ε, και πολλοί λέγανε πώς μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σφάλμα μια γυναίκα. Αλλά σχεδόν καθόλου δεν μιλάμε για την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι οι άντρες είναι, ο άντρας γενικά είναι τόσο ανεύθυνος που γονιμοποιεί τη γυναίκα ακόμα και αν δεν θέλει αυτό το παιδί. Πώς μπορεί να είναι κάποιο τόσο ανεύθυνος ώστε να αφήσει, να καταστήσει έγκυο μια γυναίκα χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του. Αλλά και σε άλλες ε, περιπτώσει. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, την βία κατά των γυναικών. Πολύ συχνά επιρρύπτουμε τις ευθύνες ε, στις γυναίκες. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Γιατί αυτή η γυναίκα δεν φεύγει από αυτή την κατάσταση. Why doesn't she just leave? Γιατί δεν φεύγει λοιπόν, δεν αποχωρεί. Αντί να θέσουμε το αντίθετο ερώτημα. Πώς γίνεται κάποιος ε, να ασκεί τέτοια βία κατά μιας γυναίκας. Να, να δώσουμε την έμφαση σε αυτόν που κάνει αυτή την ε, κολάσιμη πράξη. Και εδώ επιτέλους αυτή την έκθεση δίνουμε έμφαση στον ρόλο του άντρα και όχι στον ρόλο της γυναίκας. Ο άντρας εδώ αποφασίζει, έχει αυτό το δικαίωμα γιατί η κοινωνία του το επιτρέπει. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει το δικαίωμα να θεωρεί τη γυναίκα ως ε, αντικείμενο. Με χρηματικό αντίτιμο, γιατί μπορεί με χρήματα, με ένα ε, τέτοιο αντίτιμο, να αγοράσει ε, μια γυναίκα, λες και είναι ένα αντικείμενο. Μπορεί να ρωτήσει το όνομά της ή όχι, ανάλογα με το τι θέλει. Να ρωτήσει, δεν ρωτάει αν θέλει να είναι εκεί ή αν είναι αναγκασμένη αυτή η γυναίκα να βρίσκεται εκεί και να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί δεν έχει χρήματα να ζει στα παιδιά της γιατί ε, ήταν ε, θύμα σεξουαλικής βίας ε, κατά την παιδική της ηλικία. Κανένας δεν ρωτάει αυτή τη γυναίκα τι της συμβαίνει. Ή μπορεί να τη ρωτήσει αν το επιθυμεί, αλλά τέλος πάντων είναι επιλογή του άντρα. Είναι πολύ σημαντικό που επιτέλους δίνουμε έμφαση στον ρόλο του άντρα αντί για τον ρόλο της γυναίκας εδώ. Και μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή. Το λεγόμενο σύνδρομο της ε, Παναγίας και της ε, Πόρνης. Madonna and the Whore. Παραδοσιακά πάντα τις γυναίκες τις παρουσιάζουμε με δύο διαφορετικούς ε, τρόπους. Έχω, λέει ο άντρας, τη, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου, αυτή που είναι υπεύθυνη για την κοινωνική μου ζωή και υπάρχει και η άλλη γυναίκα, η πόρνη, που είναι το σεξουαλικό μου αντικείμενο. Δεν μπορούμε να έχουμε υπεύθυνε σχέσεις ανάμεσα σε ένα ζευγάρι όταν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο τύπων γυναικών. Όταν δεν μπορούμε να συνδέσουμε διαφορετικές ιδιότητες ε, στην ίδια γυναίκα. Πρέπει επιτέλους ε, να δώσουμε ένα τέλος ε, σε αυτό το διαχωρισμό. Κάτι ακόμα. Τι ακριβώς πιστεύουμε για αυτό το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής. Συχνά θεωρούμε, όταν μιλάμε για ελεύθερη επιλογή, ότι μπορεί κάποιος να έχει απόλυτο έλεγχο επί του σώματός του. Μπορεί κάποιος να πουλήσει ε, τα οργανά του, τα νεφρά του. Ή ας πούμε ε, υπάρχει και μια αντίστοιχη περίπτωση σε κάπου σε μια αγορά ή σε ένα πανηγύρι μπορούμε να πληρώσουμε κάποιον για να του πετάξουμε αντικείμενα. Μάλιστα αυτό ήταν ε, ε, περίπτωση υπόθεση στην νομολογία της Γαλλίας και ως δεδικασμένο έχουμε πλέον ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το σώμα κάποιου ως αντικείμενο. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα ηθικών αξιών. Μέχρι πού μπορούμε να πάμε λέγοντας ότι υπάρχει ελεύθερη επιλογή του καθένα ε, σε ό,τι φορά το σώμα του. Εγώ θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος ε, γεννιέται με μία με ένα πεπρωμένο, μια μοίρα και κάθε ανθρώπινο έχει μια αποστολή. Και όπως είπε η συγγήτρια, κανένας δεν έρχεται στον κόσμο για να αγοράζουν το κορμί του 15-20 άντρες την ημέρα. Είμαστε προορισμένοι για ανώτερα πράγματα. Γι' αυτό στηρίζω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Next is uh, please. Ευχαριστώ, την κυρία Σούμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης και οι συμβιβαστικές τροπολογίες που παρουσιάστηκαν οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση για να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών και για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, θα υποστηρίξουμε όχι όλες ε, την πλειονότητα των τροπολογιών. Και αν δεν υπάρχει κάποια τροπολογία που να είναι σε απόλυτη αντίθεση με την αντίληψη που έχουμε εμείς για το θέμα της πορνείας ε, και τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και των ανθρώπων, γενικότερα εμείς θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ε, πολύ επικοδομητική αυτή η εργασία. Και για να μην επαναλαμβάνω τώρα εδώ μία συζήτηση που αντικατοπτρίζεται στις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Ήθελα απλώς να πω ότι εμείς δεν θεωρούμε και δεν δεχόμαστε η πορνεία να θεωρείται ή να εξισώνεται με μια υπηρεσία ή με μια δουλειά. Για μας ένα επάγγελμα είναι κάτι που συνεισφέρει στην κοινωνία και στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Είναι κάτι που υλοποιεί ο άνθρωπος και συνεισφέρει στην ευτυχία του. Και δεν ε, πιστεύουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα κάτι που είναι κατάφορα αντίθετα στα δικαιώματα των ανθρώπων κατά της ύπαρξής τους. Δεν θεωρούμε ότι είναι αξιοπροπές, να θεωρούμε ότι το σώμα ενός ανθρώπου, αλλά και όχι μόνο το σώμα, αλλά και τα ιδιαίτερα στοιχεία του μπορούν να θεωρηθούν ως εμπόρευμα. Έτσι λοιπόν έχουμε κατά νου το ζήτημα αυτό. Για μας δεν υπάρχει αξιοπρεπής ε, κοινωνία. Και δεν ε, θεωρούμε ότι μπορεί ένα άτομο να αγοράζεται και να πουλιέται. Και επομένως πιστεύουμε ότι Όλες οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετικές και πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει σημαντική βαρύτητα η έκθεση αυτή στο να αλλάξουν οι δημόσιες πολιτικές σε σχέση με το θέμα της επίτευξης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Και Κυρία Ζαμπόσκα, η κυρία Νίμπλε, θέλω να το λέω, κυρία Νίμπλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που ήρθα τόσο καθυστερημένα. Είχα την ε, ε αντιπροσωπεία μου η οποία ασχολείται με θέματα δικαίου στον αραβικό χώρο που έπρεπε να προεδρεύσω εκεί και είχαμε καλεσμένους από το, τον έξω κόσμο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει γίνει αυτή η έκθεση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Mary Hannibal, η οποία έχει συντάξει μια πολύ καλή έκθεση. Εγώ υπέβαλα ορισμένε τροπολογίε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας για τις τροπολογίες μας που θεωρώ ότι έχουν σημασία και θέλω να ζητήσω από την κυρία εισηγήτρια να έχουμε την ευκαιρία να να εκφράσω την ε, αποκλίνουσα απόψή μου για τα θέματα αυτά πριν από την ψηφοφορία. Από το 2002 έχουμε ένα από τα πιο φιλελεύθερα καθεστώτα για την πορνεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Υπό την κυβέρνηση σοσιαλιστών πρασίνων υπήρξε αυτή η απόλυτη φιλελευθερωποίηση της ε, πορνείας και θεωρήθηκε ότι είναι μια, ένα επάγγελμα όπως και άλλα επαγγέλματα Ευτυχώς η νέα κυβέρνηση τώρα έχει αντιδράσει και στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει πανεπεξεργασία αυτού του φιλελεύθερου καθεστώτος αλλά θα ήθελα την κατανόηση των συναδέλφων γιατί ξέρετε ότι στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετική κατάσταση από τα άλλα κράτη-μέλη και θα ήθελα να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής πορνείας και πορνείας ως επάγγελμα να γίνεται μια διάκριση γιατί είναι αυτό ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τις εφημερίδες και τα κανάλια. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτη απαγόρευση της πονίας και εκεί υπήρξε δημόσια εξέγερση. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντιπαράθεση στο θέμα αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να επιβάλλουμε μια στάση υπεραπόλυτης απαγόρευσης. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει απαγόρευση πορνείας σε όλα τα κράτη-μέλη, αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο μαύρη αγορά και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ενώ αντίθετα αυτό το οποίο βλέπω να υπάρχει σε αυτή την καλή έκθεση της κυρίας ε, Χάνεμπολ ναι, είναι να υπάρξει μια πιο στοχευμένη στάση για τις ε, ποινικές κυρώσεις και ιδίως στα θέματα της ε, πορνείας η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνονται από την έκθεση είναι πολύ καλύτερα από το να πει κανείς ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη εξάλληψη και θέση σε παρανομία της ε, πορνείας. Μια τελευταία παρατήρηση. Πολύ σωστά η κυρία Μορβάη ανέφερε μέχρι πού φτάνει το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Αυτό είναι το αποφασιστικό θέμα. Αλλά εδώ είχαμε και σε άλλες ε, συζητήσεις το θέμα αυτό το οποίο αναφέρθηκε όταν μιλάμε για την ε, προστασία των ε, αγέννητων παιδιών. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα με το οποίο αντιμετωπίζει η γυναίκα και είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορεί κανείς να ακολουθήσει την άποψη ότι μόνο η γυναίκα είναι αρμόδια να αποφασίσει. Η άλλη άποψη είναι ότι μια γυναίκα θα πρέπει να προστατεύεται και από τον εαυτό της εάν η ελευθερία της την οδηγεί στην πορνεία και γι' αυτό η πρότασή μου, η αίτησή μου είναι ότι εγώ δεν θέλω να κρατήσω μια στάση αποχής. Στο τέλος θα την υποστηρίξω την εισηγήτρια γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό ε, σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα όμως και στην ψηφοφορία να κάνω αυτή την ε, θέση μου σαφή ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής πορνείας και εθελοντικής πορνείας και γι' αυτό έχω καταθέσει τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και η κυρία Ινφελ των Φιλελευθέρων. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάρω την πλειοψηφία, αλλά ήθελα ακριβώς να εκφράσω σαφώς αυτή τη θέση μου και θα μου βοηθήσει αυτό να υποστηρίξω την τελική έκθεση. Κανονικά εγώ δεν επιτρέπω από σε κανένα να πάρει το λόγο στις ψηφοφορίες, γιατί τώρα κάνουμε την συζήτηση και μετά γίνεται η ψηφοφορία. Μόνο η συγγήτρια, Αν θέλει να πει κάτι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, λέει κάτι. Αλλά συνήθως δεν έχουμε καμία συζήτηση πέραν διευκρινήσεων της ε, εισηγήτριας. Η συζήτηση γίνεται σήμερα. Και αυτό ισχύει για όλες τις ψηφοφορίες. Δεν κάνουμε κάποια διάκριση εδώ εναντίον σας ή εναντίον των απόψεών σας. Γενικά στις ψηφοφορίες δεν υπάρχει συζήτηση, απλώς ψηφίζουμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Δεν θέλω φυσικά να λάβω το λόγο αύριο. Απλώς θέλω να κατανοήσετε ότι οι τροπολογίες μου δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι δεν έχουν ε, λόγο ύπαρξης, ώστε το λέω αυτό για να μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση. Ναι, λέει η κυρία Χάνιμπολ, δεν θα θεωρηθούν άκυρες οι οι τροπολογίες σας το αναγνωρίζουμε αυτό. Θα υπάρχουν οι τροπολογίες σας λοιπόν προς ψήφιση αύριο. Αυτό μην ανησυχείτε. Εντάξει λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Ζαμπόσκα έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ. Και σε αυτή την νομοθετική περίοδο Αντιμετωπίσουμε και πάλι το θέμα της πορνείας. Στην προηγούμενη θητεία είχε ξεκινήσει και τότε η συζήτηση για τα θέματα αυτά. Εγώ από την αρχή να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε εσά τον ίδιο τον Πρόεδρο για την ακρόαση που οργανώσατε πριν από τα Χριστούγεννα και πρόκειται ακριβώς για το θέμα αυτό της πορνείας Υπήρξαν πολύ σημαντικοί εμπειρογνώμονες από τα κρατη που έλαβαν το λόγο για το θέμα αυτό. Ήταν όλα αυτά πάρα πολύ χρήσιμα. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, πρέπει να έχει καταρχήν μια γνώση πια για το ποια είναι η κατάσταση στην αγορά της πορνείας. Επομένως, αυτή η ακρόαση ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική για να καταλάβει κανείς την Εγώ αντιμετωπίζω αυτά τα θέματα εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω και αυτό το οποίο έχω κατανοήσει είναι ότι η αλλαγή στην προσέγγιση είναι το πιο σημαντικό θέμα. Εδώ δεν μιλάμε για την υποχρεωτική πορνεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει όλοι. Το έχουμε όλοι απορρίψει κατά 100%. Είναι περισσότερο αυτό, αυτή η λεγόμενη εθελοντικού χαρακτήρα πορνεία και υπάρχει και μια αλλαγή κλίματος και προσέγγισης όπως φάνηκε και από την ακρόαση. Και αυτά που είπε η κυρία Ζούμπερ προηγουμένως δείχνει ότι ακόμα και η νόμιμη πορνεία αντιμετωπίζεται πια με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γινόταν πριν από 10 χρόνια. Γι' αυτό θέλω εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Χάνιμπαλ γιατί είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα το οποίο έπρεπε να φέρει σε πέρας με την επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν και αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτών οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία επιτρέπουν ενώ άλλα απαγορεύουν την δραστηριότητα αυτή. Εγώ από προσωπική άποψη μπορώ να πω ότι και στην προσωπική μου ζωή και στην πολιτική μου ζωή πάντα έχω υποστηρίξει τα δικαιώματα των ε, των παιδιών. Η σοβαχική κυβέρνηση έχει περάσει ένα πάρα πολύ φιλεύθερο νόμο για την ε, εθελοντική διακοπή της κοίησης η Τσεχία έχει προχωρήσει σε μια αρκετά φιλελεύθερη νομοθεσία που έχει απλώς χρονικό περιορισμό για την άμβλωση. Εγώ πάντα όμως προσπάθησα στην πολιτική μου ζωή να έχω σαν κύριο γνώμονα την προστασία της ζωής και αυτό είναι το ίδιο πράγμα που έχει να κάνει με την πορνεία. Θέλω να προασπιστεί η προσωπική αξία και αξιοπρέπεια και αυτό αποτελεί για μένα ένα πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να τύχει προστασίας. Κατανοώ αυτά που λένε οι συνάδελφοι που αναφέρονται στα θέματα της ε, εθνικής ρύθμισης και της επικουρικότητας. Και ως ε, σκιώδης εισηγητρία θέλω να σας πω ότι το ΕΛΚ θα υποστηρίξει τις συμβαστικές τροπολογίες και σε πολλά σημεία θα ζητήσουμε χωριστές ψηφοφορίες. Σε άλλες περιπτώσεις θα κρατήσουμε μια στάση κατά συνείδηση ψηφοφορίας γιατί είναι πάρα πολλά τα καθεστώτα και οι νομοθεσίες που ε, διαφέρουν στα κράτη-μέλη μας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσει να γίνει δεκτή αυτή η έκθεση μετά από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και η έγκριση αυτής της έκθεσης θα είναι ένα πολύ καλό μήνυμα από τη δική μας Επιτροπή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναδίνω το, λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα εγώ εδώ. Ευχαριστώ. Τα δέκα χρόνια που έχω διανύσει εδώ, συζητάμε κάθε χρόνο αυτό το θέμα, ή αν όχι κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο και δημιουργεί ε, διάφορες αντιπαραθέσεις, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν και κάποια πολύ μεγάλα σημεία συμφωνίας και πρέπει να το επενθυμίσουμε αυτό. Πάντοτε υπάρχουν κάποιες πτυχές ε, επί των οποίων αν δεν υπάρχει ομοφωνία υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία και είναι πτυχές που μπορούμε να βελτιώσουμε. Εμπορία ανθρώπων προφανώς που δεν σχετίζεται μόνο με την πορνεία αλλά και με άλλες πτυχές. Κάποιοι άνθρωποι καταλήγουν στην πορνεία και πρέπει όχι μόνο να το καταδικάσουμε αλλά και να το διώκουμε με κάθε μέσο για την παιδική πορνεία όλοι συμφωνούμε ότι δεν δεχόμαστε ε, καθόλου την ύπαρξη τέτοιων συζητημάτων ε, και επιμένω είπα ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που επίσης έχουν να κάνουν με τη χρήση παιδιών ε, για άλλους σκοπούς και δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε και το θέμα της εξαναγκαστικής πορνείας. Συμφωνώ με την κυρία Νίμπλερ ε, και στην προηγούμενη θητεία την κυρία Σαβόρσκα ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Κάναμε διάφορες κοινέ δράσεις για να καταγγείλουμε την εξαναγκαστική πορνεία. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για να κάνουμε μια δουλειά από κοινού. Υπάρχουν πάντως και άλλες πτυχές και δυστυχώς ε, η κυρία Λούνατσεκ σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά ε, υπάρχουν ε, κάποια σχόλια δικά της και υπάρχουν κάποιες πτυχές που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να καθορίσω τις θετικές πτυχές ορισμένων μέτρων. Παραδείγματος χάρη, απόλυτη απαγόρευση της πορνείας. Δεν ξέρω. Και έχω κάποιες αμφιβολίες. έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα είναι αποτελεσματική για να αφαιρέσει κινήτρα από την προσφυγή στην ε, πορνεία. Και βασίζομαι στην εμπειρία που είχαμε σε πολλές χώρες. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση και βάσει της εμπειρίας που έχουμε, ότι αν έχουμε ένα πλαίσιο με σαφείς κανόνες και που να εγγυάται ότι υπάρχουν κάποιες νομικές απαιτήσεις και ε, να μπορούν ε, οι άνθρωποι να προσφεύγουν στον νόμο και να υπάρχει ασφαλεία δικαίου, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί οι ορισμένοι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα να εγκαταλείψουν αυτή τη δραστηριότητα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα μπορέσουμε να διώκουμε καλύτερα ε, κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες. Δηλαδή ε, να μην ε, προσπαθήσουμε να κρύψουμε μια πραγματικότητα που υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω μιας απαγόρευσης γιατί ακόμη και αν την απαγορεύσουμε θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε ένα σαφές ε, πλαίσιο αδιαφεσβήτητο που να επιτρέπει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο να διώκουμε την εμπορία ανθρώπων, την εξαναγκαστική πορνεία, την χρησιμοποίηση παιδιών και φυσικά οποιοδήποτε άλλο έγκλημα που σχετίζεται με αυτές τις πρακτικές. Αυτό από τη μία πλευρά και το λέω γιατί από τη σκοπιά των πρακτικών που έχουμε στην Ευρώπη έχουμε διάφορα μοντέλα και ορισμένα είναι πολύ αποτελεσματικά για κάποια πράγματα και άλλα για κάποια άλλα. Εγώ στην περίπτωση αυτή ότι ε, εγώ δεν τα έχω ξεκαθαρισμένα τα πράγματα, δηλαδή ακόμη και αν ε, ποινικοποιήσουμε τον πελάτη. Δεν είμαι σίγουρος ότι ε, θα αφαιρέσουμε όλα τα κίνητρα και Επίσης, ε, το να, αν και δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε τους ανθρώπους που επιδίδονται στις δραστηριότητες αυτές, το γεγονός ότι ποινικοποιείται η δραστηριότητά τους έμεσα θέτει και τους ανθρώπους αυτούς σε κατάσταση κινδύνου. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι από τη σκοπιά της νομιμότητας της δραστηριότητας ε, ορισμένοι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κρυσόπους οργανώσεων και στην Ισπανία έχουμε μιλήσει με πολλές οργανώσεις γυναικών ε, βασικά γυναικών, αλλά υπάρχουν και άνδρες ε, που είναι εργάτες του σεξ και επομένως από τη σκοπιά του πετερνολισμού αυτό μου θέτει ένα πρόβλημα Δηλαδή το να μπω εγώ σε κατάσταση να αποφασίσω για το αν είναι ή δεν είναι αξιοπρεπές. Υπάρχουν πάρα πολλέ ε, δουλειές που δεν είναι αξιοπρεπείς και εδώ έχω τις αμφιβολίες μου για το αν ε, έχουμε ή δεν έχουμε την υποχρέωση να στιγματίσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη δραστηριότητα. Και το λέω σε εμφωλία, γιατί αν ακούσει κανείς τις οργανώσεις γυναικών που εργάζονται στον κλάδο, Υπάρχουν διάφορες επόψεις ε, που και αυτές είναι αποδεκτές όπως άλλες και εγώ νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να στιγματίζουμε τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, τελικά θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Νίμπλερ, δηλαδή να ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να επιτρέψουμε και να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση Βασικά γιατί δεν βρισκόμαστε ενώπιον ενός θέματος που απλώς με μια απαγόρευση θα επιληθεί εν μια νυχτή. Και μια τελευταία σκέψη. Από τη σκοπιά του να μπορούμε να εγγυθούμε τα δικαιώματα των γυναικών που μπαίνουν στα δίκτυα αυτά, το γεγονός του να καταστήσουμε ορατή αυτή τη δραστηριότητα είναι μια οδός πολύ πιο ασφαλής για τα άτομα αυτά για να μπορούν να προστατεύονται περισσότερο τα δικαιώματά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βοηθηθούν και να εγκαταλείψουν αυτή τη δραστηριότητα. Ξέρω ότι είναι μια συζήτηση πολύ παθιασμένη, προκαλεί τα πάθη, πολλά έτη τη συζητούμε θα συζητούμε τα θέματα αυτά και φυσικά και η δική μου θέση έχει εξελιχθεί ανάλογα με τη συζήτηση. Όμως, μου προκαλεί κάποιο φόβο το σημερινό κείμενο της έκθεσης. Νομίζω ότι πηγαίνει υπερβολικά προς μία γραμμή που είναι σκανδιναβική, το σκανδιναβικό μοντέλο και δεν ξέρω αν είναι το πρέπον. Επί της αρχής νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κύριο Γκούσταυσον ότι υπάρχει πολύ περιθώριο για να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών και τις συνθήκες στις οποίες, ζουν. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, τέτοιες ε, καταστάσεις ε, που πραγματικά ζημιώνουν και τα άτομα αλλά και τις κοινωνίες. Ευχαριστώ. Πρέπει να συμφωνήσουμε για όλα, αυτό είναι αλήθεια αλλά για πολλά συμφωνούμε. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Τότε να δώσουμε και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Κυρία Χάνιμπομ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση που ήταν ε, πραγματικά μια πολύ επικατομματική συζήτηση και καταφέραμε να διαφωνήσουμε με έναν ε, πολύ θετικό τρόπο και σας ευχαριστώ γιατί και το 2002 το είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή και δεν ήταν έτσι η συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους ε, από καρδιάς για τον τρόπο που του χειριστήκατε το θέμα αυτό και τις επικοδοματικές σας προτάσεις. Ανέκυψαν πολλά ζητήματα από την ε, κουβέντα. Θα ήθελα να ξεκινήσω την κυρία Νίγκερ και Ζαμπόσκα. Κυρία Νίμπλερ πρώτα, γιατί μιλήσατε πρώτη. Ε, για την εξαναγκαστική πορνεία. Ξέρω ότι διαφωνούμε και σέβομαι τα όσα είπατε για τη Γερμανία και τη θέση της Γερμανίας, πώς θα άλλες δηλαδή κατά της Γερμανίας αν προσέγγιση έχετε καταθέσει τροπολογίε ε, που κάνουν λόγο για εξαναγκαστική πορνεία και πορνεία. Μπορώ να τις αποδεχθώ όταν όμως μιλάμε εν γέννη για την πορνεία. Γιατί εγώ είμαι κατά και των δύο. Θα τις στηρίξω λοιπόν αυτές τις τροπολογίες και έτσι φαντάζομαι απαντώ το βασικό σας ερώτημα. Παρότι καλό ε, για υιοθέτηση του ειδικού μοντέλου, βεβαίω δεν θα ήθελα να το επιβάλλω στα κρατημέλη έτσι. Εντάξει, βεβαίως δεν είναι μια νομοθετική πρόταση, είναι μια ε, έκθεση πρωτοβουλία ε, με στόχο να αναλύσουμε την κατάσταση και να βρούμε λύσεις ε, γιατί είναι σημαντικό σε τέτοιου είδου εκθέσει να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Και έτσι απαντώ ε, στην πατρίστη του κ. Βέβερ. Επιλέγω μία προσέγγιση, μία γραμμή, γιατί εγώ θεώρησα ότι αν έπρεπε να κάνω τέτοια έκθεση, θα έπρεπε να καταλήξω σε συγκεκριμένες προτάσεις. Γι' αυτό και τα έχω εξετάσει πολύ προσεκτικά και γι' αυτό συστήνω το σουηδικό ε, πρότυπο. Το οποίο δεν απαγορεύει ουσιαστικά την, απαγο... την ε, πορνεία. Κάποιοι ανέφεραν την απαγόρευση της πορνείας. Η ποινικοποίηση του αγοραστή δεν σημαίνει και απαγόρευση της πορνείας. Απλώς ε, καθιστά ποινικό αδίκημα την αγορά τέτοιων υπηρεσιών. Το μοναδικό κανονιστικό πλαίσιο ε, είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της πορνείας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι η λύση που πρέπει να επιλέξουμε. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Η νομιμοποίηση της πορ... και η ποινικοποίηση της πόρνης αλλά και της ε, ε, λειτουργίας ε, ενός ε, Πορνίου δεν έχει οδηγήσει τέτοια αποτελέσματα. Μόνο με αυτό το μοντέλο μπορούμε να οδηγήσουμε στην μείωση της ε, ζήτησης. Και αυτό εγώ συνιστώ είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να κινηθούμε προς ε, την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Και εδώ δεν θέλουμε να στιγματίσουμε για να ε, κατακρίνουμε τις γυναίκες που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Στόχο μα είναι να μιλήσουμε εδώ για την ισότητα των φύλων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εγώ είμαι κατά τη πορνεία γιατί θεωρώ ότι ε, πλήττει την ισότητα των φύλων. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε, όχι τους εργαζομένους του ίδιου. Ήμουν αρκετά σαφή στην έκθεση και θα υποστηρίξω όλες τις τροπολογίε που στηρίζουν τις γυναίκες που θέλουν να φύγουν. Και υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε από αυτού. Αλλά και για το ασφαλές περιβάλλον. Όπως είπα και εισαγωγικά, δεν νομίζω ότι κάποια γυναίκα επιλέγει την πορνεία. Το κάνουν εξαιτία διαφόρων αιτιών, οικονομικών δυσχεριών ή σεξουαλική βία που έχουν βιώσει ε, στην παιδική τους ηλικία, παιδοφιλία και το καθεξής. Δεν είναι λοιπόν ελεύθερη επιλογή και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι περισσότερες ε, πόρνες θέλουν να ξεφύγουν από την πορνεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ε, που να τις στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνώ λοιπόν και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε ε, τις γυναίκες που θέλουν να ξεφύγουν από την πορνεία και να τις βοηθήσουμε να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Δεν πρόκειται για στιγματισμό. Ελπίζω κύριε Νίπλερ έτσι να απάντησα στα δικά σας σχόλια. Κυρία Σαπούσκα, χαίρομαι ιδιαίτερα που το ΕΛΚ, ελπίζω κιόλας να με στηρίξετε, είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Και ήδη υπάρχει συνένεση επί της βάσης. Μπορεί να διαφέρουμε σε ό,τι φορά τις λύσεις. Αλλά στα βασικά όλοι συμφωνούμε. Δύο πράγματα ακόμα για τα ανήλικα άτομα. Ξέρω ότι χρησιμοποίησα εκτεταμένα τον όρο κορίτσια στην έκθεσή μου. Ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, διαφορετικές ηλικίες ε, συνένεσης. Αλλού έχουμε 21, στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 16. Βεβαίω, με τα χαρά να βρούμε έναν όρο που να καλύπτει όλα τα κρατη γιατί βεβαίως θέλουμε να δώσουμε απόλυτη προστασία ε, στα ανήλικα κορίτσια και δεν υπάρχει ε, εκεί βεβαίως ε, καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα όταν πρόκειται για ανήλικες. Μετά, για τον ποινικό χαρακτήρα θα πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε, όπως επεσήμεναν πολύ ότι ε, υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος πίσω την πορνεία. Όλο αυτό το δίκτυο θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Αν ε, μειώσουμε την ζήτηση, βεβαίως θα μειωθεί και ολόκληρος αυτός ο τομέας. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που ήθελα να θίξω. Όπω είπα και προηγουμένως, χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε μια τόσο επικοινωνική συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπω ε, είπε και η συγγήτρια, η συζήτηση ήταν πολύ καλή. Τα έχουμε συζητήσει επί μακρόν όλα αυτά. Θα ψηφίσουμε αύριο και θα πάει το θέμα στην ψηφοφορία στην δεύτερη από τις Ολομέλειες του Φεβρουαρίου. Κλείνουμε εδώ λοιπόν αυτό το σημείο της μέσας διάταξης και τώρα περνάμε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Κλείνουμε εδώ λοιπόν την πρωινή συνεδρίαση. Και... Ουσιαστικά στις 11.30 πρέπει να ξεκινήσει ε, η συνεδρίαση των συντονιστών. Αλλά από ό,τι βλέπω είμαστε όλοι εδώ, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως. Uh, exactly.